για την αναβολή της ψηφοφορίας αυτού του ψηφίσματος ήταν σοφή. Αύριο θα εγκρίνουμε μια πληρέστατη έκθεση που θα είναι χρήσιμη και για την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε. Ο, κύριος Στογιάννοφ έχει το λόγο.